Α, αλλά θα συνεχίσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου και ας ελπίσουμε ότι οι συνάδελφοι που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση να ε, βγουν ήσυχα από την αίθουσα και ευχαριστώ τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας και παρακολούθησε τις συζητήσεις μας. Συνοχή. Colleghi, iniziamo Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Έχω διάφορες αιτήσει για παρεμβάσεις. Μπορούμε λοιπόν ε, να δουλέψουμε μόνο μέχρι τις 3 ε, παρατέταρτο. Και αυτό για να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να προετοιμάσουν ε, την αίθουσα που θα ε, ξαναξεκινήσει ολομέλεια στις 3. Άρα δηλαδή οι υπόλοιπες επεξηγήσεις ψήφου που δεν θα μπορέσουν να γίνουν σήμερα θα εξεταστούν αύριο. Και άλλες επεξηγήσεις ψήφου, ψήφου μπορούν να κατατεθούν ε, γραπτός. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα των ε, Ολομελιών για το 2016 και ζήτησε το λόγο για επεξήγηση ψήφου ο κύριος Ντάνιελ Ανάν. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Τιπρέοδρε. Όλοι γνωρίζουμε τα επιχειρήματα κατά της μετακίνησης αυτής από Βρυξέλλες σε Στρασβούργο. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω τα επιχειρήματα. Αυτή η συνάντηση συμβολίζει την ακινησία και την αντίσταση στην αλλαγή για να αποφύγουμε την γραφειοκρατία. Θυμηθείτε αυτό που είπε και ο Φρίτμαν, θυμηθείτε τι γίνεται έξω από τα γραφεία μας, πόσο πολύ αντιστεκόμαστε Υπάρχει όμως ο κλάδος της μεταφοράς, μεταφερόμαστε εδώ και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά υπάρχει για να εξασφαλίσει τους ίδιους της τους υπαλλήλους και τίποτα άλλο. Στην πρακτική αυτό είναι αδύνατον να υπάρξει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση υπέρ των Βρυξελών. Είναι η τυραννία των χωρών μελών. Γιατί το κάνουν αυτό, οι κυβερνήσεις δεν έχουν καμία φιλοδοξία. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και αν λένε οι πολίτες μας και πιστεύουν, το σύστημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει προς όφελος των τυχερών που απασχολούνται μέσα σε αυτό το σύστημα εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Χάναν. Περνάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση ε, για τη σύσταση ε, σχετικά με τις ε, δυνατότητες που μπορεί κανείς ε, να εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση της, ε, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα στηρίξω την πρόταση αυτή, η οποία ρυθμίζει τα θέματα νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, στην Τσεχία. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένο που η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει τις ε, ανώνυμες μετοχές και πρέπει να γνωρίζουμε ποιος, σε ποιον ανήκουν τελικά διάφορες επιχειρήσεις. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί πολύ στην ε, Τσεχία και έχουμε προτείνει να καταργηθούν οι ανώνυμες μετοχές. Είμαστε στον καλό δρόμο και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε τον ίδιο δρόμο γιατί οι ανώνυμες μετοχές επιτρέπουν νομιμοποίηση παράνομου χρήματος και παράνομων κεφαλαίων και μπορεί να πρόκειται και για ε, τρομοκρατικές δραστηριότητες. Είναι σωστή λοιπόν τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα την τρομοκρατία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Τζιλ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί δίδει σημαντικά εργαλεία για την αποφυγή της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και μπορεί να παίξει και σημαντικό ρόλο ε, στην ε, μείωση των χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όσο πιο διαφανές είναι το σύστημα τόσο το καλύτερο. Με την δημόσια καταχώρηση νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις ροές. Όμως όπως δείχνουν τα πρόσφατα φορολογικά σκάνδαλα εξαρτώμεθα κατά πολύ από τις προφορίες που δίδουν οι εργαζόμενοι ε, εσωτερικά στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε ε, και στην συνεργασία των κρατών μελών που πολλές φορές δεν θέλουν να το κάνουν. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο λοιπόν για την προστασία των ε, πληροφοριοδοτών. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Ανάν για ένα λεπτό. Παρατήρησα ότι οποτεδήποτε κάποιος θέλει να διευρύνει τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, Europol, Eurojust κλπ. Χρησιμοποιούν πάντοτε το επιχείρημα της ασφάλειας. Γιατί η ασφάλεια υποτίθεται ότι είναι αχτύπητο επιχείρημα. Τι έγινε με το FBI στην Βόρεια Αμερική. Το FBI ακριβώς δρά, όπως ακριβώς αναφέρει αυτή η έκθεση εναντίον του ξεπλήματος χρήματος, της τρομοκρατίας κλπ. Και τι έγινε. Έγινε ομοσπονδιακή αστυνομία για όλες τις ΗΠΑ τελικά. Ε, παρόλο ότι ε, μάλλον ε, ε, αισθανόμαστε και λιγότερο ελεύθεροι και όχι περισσότερο ασφαλείς ε, χωρώντας τέτοιου αρμοδιότητες και όχι μόνο σε αυτό το θέμα αλλά και σε πολλά άλλα θέματα γεωργικής πολιτικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ. Έχουμε υπηρεσίες ε, πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει σε εθελοντική βάση να συνεργάζονται μεταξύ τους. Η ανάγκη έχει αποδειχθεί ότι είναι η ε, δικαιολογία για οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριο Φλάνναγκαν. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Δεδομένη τη εμπειρία τη Ιρλανδία από την τρομοκρατία και από την κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο και πώ αυτό χρησιμοποιείται για την νομοποίηση παράνομου χρήματο και χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ όλου του Ιρλανδού. Δεν χρειάζεται να σα πω τώρα πώ η τρομοκρατία έπληξε την Ιρλανδία για χρόνια. Υπάρχουν πολλοί οποίοι δεν έχουν ακόμα δικαιωθεί. Όμω τα αποτελέσματα είναι άλλο είδου τρομοκρατία. Είναι μια τρομοκρατία πιο ευρέω διαδεδομένη και ενδυμική Μιλάω για την ε, πιστοτική τρομοκρατία που επιβάλλεται στους ανθρώπους ολόκληρο τον κόσμο δυσανάλογα από συμφέροντα των οποίων ε, οι δράσεις διευκολύνονται από κυβερνήσεις. Η ίδια η δικιά μας κυβέρνηση στην Ιρλανδία για παράδειγμα, η οποία τελικά είναι όμοιρος του φύση και είναι τα ίδια οικονομικά συστήματα τα οποία ε, οδηγούν τον κόσμο σε εξάρτηση και οι New York Times έχουν ε, αναφερθεί στο Far West ε, το οικονομικό. Η ιδέα λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι ε, θα έπρεπε, αλλά όχι η ίδια να εφαρμόζει τέτοια οικονομική τρομοκρατία, γιατί τελικά είναι περίπου ανέκδοτο το ότι μπορεί να μας προστατεύσει. Ευχαριστούμε κύριο Σόγκορα, ένα λεπτό. Είμαι υπέρ της οδηγίας αυτής κατά της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και νέε απειλέ. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να πάμε και ακόμα πιο μακριά από τις συστάσεις που έκανε το 2012 η Task Force για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο προστασίας με υψηλές προδιαγραφές. Η κατάχρηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων χρηματοδοτεί τελικά ε, τρομοκρατικές δράσεις και πλήττει την σταθερότητα του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια συνολική αντίδραση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάρ έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένας φιλόσοφος είχε πει κάποτε ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην ροή των πραγμάτων. Βεβαίως και Θέλουμε εκείνη η αγορά και πρέπει να μεριμνήσουμε οι άνθρωποι να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη και θέλουμε να πλουστεύσουμε τις χρηματοπιστωτικές ροές. Αλλά δυστυχώ βεβαίω σε τέτοιου είδου εξελίξει προκύπτουν και αρνητικέ εξελίξει, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, ε, ε, χρηματοψηφιακή τρομοκρατία. Πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρόσθετα με την υπάρχουσα πρόταση η Κομισιόν κατέθεσε και άλλε προτάσει. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να παρακαλέσω για το εξή. Αυτή την τέταρτη οδηγία περί ξεπλήματο βρώμικου χρήματο πρέπει να την παρακολουθήσουμε διότι μερικές φορές ε, το κακό, το αρνητικό έχει πολύ μεγάλη φαντασία και εμείς δεν πρέπει να αποκλίνουμε από την ύπαρξη των προβλημάτων. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πέτυρ, για... η κυρία Πέτυρ, με συγχωρείτε, για ένα λεπτό. Ε, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την πρόληψη της νομοποίησης ε, ε, παρανομών εσόδων ε, και για προκειμένου επίσης να παρεμποδίσουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις δεδομένων των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα γύρω από την Ευρώπη είμαι υπέρ τέτοιων μέτρων που βοηθούν το σύστημα να κατασταθεί πιο διαφανές. Επίσης στηρίζω την διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών με την καταγραφή ε, σε κεντρικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη όλων των ονομάτων ε, ε, των δικαιούχων των μετόχων με προφανώς με τις κατάλληλες δίτες προστασίας. Ευχαριστούμε κύριε Πετήρ, ο κύριος Γκόλνης. Η καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος και άρα καταπολέμηση της οργανωμένης τρομοκρατίας, ναι. Αλλά πιστεύετε σοβαρά ότι το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία περνάνε από τα συνηθισμένα κυκλώματα, τα τραπεζικά. Μα το σύστημα λειτουργεί ανώμαλη στην ίδια τη δικιά μου τη χώρα, στη Γαλλία. Χάρη στην ρύθμιση που έχουμε, κάθε τραπεζίτης καταλήγει να είναι κατάσκοπος ο οποίος ε, προσπαθεί να κατασκοπεύσει τους πελάτες τους. Έτσι πριν από λίγο καιρό για να πληρώσουμε 10.000 ευρώ που ήταν ε, μια πίστοση που είχα στο λογαριασμό μου έπρεπε να δικαιολογηθώ στην τράπεζό μου η οποία με έψαξε, βρήκε περίεργη την ε, συναλλαγή μου και με ρώταγε γιατί τα κάνω. Εγώ του είπα ότι τι να κάνουμε, οι μετρέσεις σήμερα κοστίζουν πιο ακριβά από ό,τι παλιότερα. Δεν ικανοποιήθηκε όμως ο τραπεζίτης μου από αυτό, οπότε τελικά ενημερώνουμε την οικονομική αστυνομία, γίνονται έρευνες, μα αυτά είναι τελείως ανώμαλα πράγματα από την ομοθεσία αυτή. Όπως το διαπιστώνουμε και στην ε, Credit Bank, την ίδια τη τράπεζα που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν τους φτάνει το διαβατήριό σας το ευρωπαϊκό για να δικαιολογήσετε τον τόπο κατοικία σας. Αυτή είναι τρομοκρατία οικονομική η κυρία Ιβάνα Μάλετιτς για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της ε, πρόληψης ε, της ε, νομοποίησης εσόδων, από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντικό για όλα τα κρατημέλη γιατί διαφορετικά τα χρηματοπιστωτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θα υποστούν πλήγμα. Ε, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας εναντίον αυτών των δραστηριοτήτων. Στηρίζω τις τροποποίησεις οδηγίας όπου προτείνεται, προτείνονται, προτείνεται να δίδονται διάφορα στοιχεία προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες. Και επίσης προτείνεται κάθε 6 μήνες να γίνεται ανάλυση κινδύνου. δίδεται ιδιαίτερο βάρος στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά. Τελείωσε λοιπόν η συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό για την ομοποίηση εσώτων από παράνομες ε, δραστηριότητες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις επεξηγήσεις ψήφου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές ε, χρηματικών ποσών. Και έχουν ζητήσει το λόγο ο κύριος ε, Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και το σχέδιο αυτό και το προηγούμενο και τροποποίηση της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει σαν σκοπό να συγκεντρώνονται περισσότερες πληροφορίες όταν γίνονται μεταφορές χρημάτων. Ε, φυσικά και συγκέντρωση αυτή πληροφοριών θα έχει σαν αποτέλεσμα οι πολίτες να νομίζουν ότι συγκεντρώνουμε πληροφορίες ε, που τους αφορούν και που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τους βίο. Η διεθνής τρομοκρατία από την άλλη μεριά χρηματοδοτείται με χρήματα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να έχουμε τις πληροφορίες αυτές και να τις χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ε, δραστηριοτήτων. Είμαι υπέρ του σχεδίου αυτού, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει έρευνα για μια ύποπτη συμπεριφορά, αν υπάρχει κάποια υπόνοια δηλαδή για σοβαρή και σοβαρό έγκλημα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τζίλ έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ κυρία Τζίλ. Ευχαριστώ. Στήριξα την ρύθμιση αυτή όσον αφορά την μεταφορά ε, χρηματικών ποσών. Πρέπει να έχουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και καλύτερη προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς που καταγγέλουν πρακτικές ε, παράνομες. Και όποτε γίνονται καταχρήσεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν και σώματα επιβολής του νόμου στις χώρες μέλου και να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Είναι απαράδεκτο πραγματικά δισεκατομμύρια ευρώ να εξακολουθούν να περνάνε και να χρησιμοποιούνται για παράνομες ενέργειες κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε κυρία Τζιλ. Το λόγο έχει η κυρία Μαλετίτς. Ένα, Ένα λεπτό κι εσείς. Ένα. Ευχαριστώ. Προκειμένου να προλάβουμε και να ερευνήσουμε την ευνομοποίηση παράνομων εσόδων. Αυτός ο κανονισμός έχει ε, στόχο να ε, βελτιώσει τον έλεγχο μας επί των μεταφορών χρηματικών ποσών, ε, αυξάνοντας τον αριθμό των εγγράφων που τις συνοδεύουν. Η νομοθεσία αυτή θα ενισχύσει το σύστημα ελέγχου και θα αυξήσει τις κυρώσεις. Ο κανονισμός αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, διότι άπτεται πληροφοριών, δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να μεταδίδονται προκειμένου να ταυτοποιούνται ε, οι συναλλασσόμενοι. Οι αλλαγές που επιφέρει είναι σημαντικές, διότι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και πολύ γρήγορα. Υπάρχουν ε, ε, καινούργια παραθυράκια τα οποία θα πρέπει να κλείσουν για να εξασφαλίσουμε και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στήριξα αυτή την σύσταση. Ευχαριστώ. E Πολύ ωραία. Και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για τη σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την αφαιρεγκαιότητα, τις διαδικασίες αφαιρεγκαιότητας. Εν τω μεταξύ θέλω να σας ε, πω ότι υπάρχουν και ακροατές ε, επισκέπτες στην αίθουσα και τους χαιρετίζω, αλλά απλά να σας πω και να σας εξηγήσω ότι εδώ δεν είναι ολομέλεια, απλά γίνονται επεξηγήσεις ψήφου. Ήδη έχουν ψηφίσει οι ευρωβουλευτές. Το λόγο λοιπόν θέλω να δώσω ε, στον κύριο Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στηρίζω την αλλαγή αυτή κανονισμού όσον αφορά τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Συμμετείχα στις συζητήσεις χτες, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα χτες να πάρω το λόγο. Γι' αυτό και ζήτησα να συμμετάσχω στις επεξηγήσεις ψήφου. Για μένα το πιο σημαντικό στον τομέα αυτό είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα μητρό αφαιρεγγιότητας Έχω ασχοληθεί πολύ με το δίκαιο φερεγκαιότητα στην Τσεχία ως θέος Υπουργός Δικαιοσύνης και γνωρίζω ότι χρειαζόμαστε δημόσιες πληροφορίες, πληροφορίες για όσους είναι αφαιρέγγοι, πληροφορίες που και διασυνοριακά πρέπει να είναι διαθέσιμες ώστε οποιαδήποτε επιχείρηση να μπορεί να ενημερωθεί για το χρέος κάποιου άλλου φορέα σε μια άλλη χώρα μέλους. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια επαναστατική αλλαγή η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες αφαιρεγκαιότητα σε όλες τις χώρες μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ευχαριστούμε κυρία Τζίλ. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί πιστεύω ότι είναι ισορροπημένη. Είναι πολύ θετικό που ενημερώνουμε την ε, νομοθεσία αυτή μετά από 10 χρόνια εφαρμογής. Ο κανονισμός καλύπτει 50.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναμειχθεί σε διαδικασίες αφαιρεγγιότητας διασυνοριακά. Πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες για τη δικαιοδοσία. Η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και ποιος είναι ο νόμος που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφές. Δεν πρέπει να υπάρχουν μικτές, επιχειρήσεις, ε, διαδικασίες. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το πρόσθετο κριτήριο των τριών μηνών προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φλάναγκαν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Μέχρι πριν από δύο χρόνια η, η Ιρλανδία είχε ένα από τα πιο αυστηρά καθεστώτα φερεγγιότητα στην Ευρώπη. Ε, με πολύ παλιά νομοθεσία. Τότε ήμουν ε, βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εξαιτία τη ε, κρίση εργαστικών δανείων η τότε κυβέρνηση που είναι και σημερινή χρειάστηκε να εισάγει πιο σύγχρονη νομοθεσία. Ε, Παρ' όλα αυτά, αντί η καινούργια νομοθεσία να είναι να ωφελήσει τον κόσμο επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από το τραπεζικό κλάδο και αυτό δυσκόλυψε πάρα πολύ αυτούς που είχαν στεγαστικά δάνεια. Τα, οι τράπεζες πήραν το δικαίωμα ε, να διαπραγματευτούν τη δυνατότητα ε, να εφαρμοστούν οι κανόνες περί ε, ε, μετά χρειάστηκε η κυβέρνηση να ξανακινηθεί, χωρίς όμως να μπορέσει να άρει τις ευλάβες που έχει δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ηρωνικό όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιούργησε την κρίση στην Ιρλανδία θα χρησιμοποιήσει, θα δημιουργήσει ε, κανόνες για να την ε, διασώσει. Ευχαριστώ. Πέτυρ. Ευχαριστούμε κύριος Πετύρ. Κύριε Πετύρ. Ευχαριστώ. Στήριξα την έκθεση αυτή και ελπίζω ότι όλες οι διαδικασίες αφαιρεγκαιότητας θα επιταχυνθούν τώρα. Ελπίζω επίσης ότι θα επηρεάζονται αρνητικά λιγότερο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες περνάνε από τέτοιες διαδικασίες. Πρόκειται για έναν εφιάλτη για κάθε επιχείρηση. Η διαδικασία αφαιρεγγιότητας είναι κάτι το οποίο ε, κρατάει χρόνια και αρχίζει μόνο όταν η διαδικασία είναι απελπιστική. Στην Κροατία υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν πολύ περίεργες συμφωνίες και ρυθμίσεις τελικά που λαμβάνουν χώρα. Δεν ξέραμε πώς θα καθοριστεί τελικά ποιος θα πρέπει να πληρωστεί. Πιστεύω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική. Χαίρομαι που εγκρίθηκε και ελπίζω ότι θα βοηθήσει να αλλάξουν τα αρνητικά στην Κροατία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Ιβάνα Μάλετιτς έχει τώρα τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαδικασίες ε, αφαιρεγγιότητας ε, διαφέρουν από κράτος σε κράτος και επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ε, όπως επίσης και τη σταθερότητα των κρατών μελών εν υπό το φως της κρίσης. Ο στόχος της, ε, ε, της αυτής ε, είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να λειτουργήσουν καλύτερα. Οι συστάσεις είναι σαφές ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι σαφείς και γρήγορες. Ε, η κρατική νομοθεσία σε αυτό τον τομέα έχει κριθεί ως μάλλον αδύναμη και η κυβέρνηση θα πρέπει να την βελτιώσει το συντομότερο δυνατό. Ο κανονισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, γι' αυτό το λόγο τον υποστήριξα. Περνάμε στην έκθεση Winkler για την αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Το λόγο έχει η κυρία Αρένα. Δεν τη βλέπω όμως εδώ. Οπότε η κυρία Τζιλ. Παρακαλώ, για ένα λεπτό κυρία Τζιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που αναβάλαμε την τελική ψηφοφορία όσον αφορά το θέμα αυτό και θα πάμε σε τριμερή διάλογο. Είμαι όμως απογοητευμένος από την θέση που υιοθέτησε το ΕΛΚΑ και το ΙΣΙΑΡ. Γιατί δεν θέλουν να υπάρχει υποχρέωση. Γνωρίζουν πολύ καλά και εκείνοι όπως και εμείς ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας, στα κομπιούτερ κτλ. Ε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα μεταλλεύματα αυτά λοιπόν, δεν τα παίρνουμε από ανθρώπους που επιτυχαίνουν κακή κακής εκμετάλλευσης. Μόνο αν υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες θα το καταφέρουμε αυτό. Ας ελέγξουν τι γίνεται σήμερα στην αλυσίδα αυτή των μεταλλευμάτων. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Τα μεταλλεύματα αυτά θα εξακολουθούν να πουλούνται στις εμπορικές αλυσίδες και θα προέρχονται κυρίως από την Κίνα είναι όλο και πιο δύσκολο να καταλάβουμε τη θέση τους, δεδομένου ότι δεν πληρώνουμε κανένα, οι επιχειρήσει δεν πληρώνουν ε, πολλά, ε, πολλά χρήματα. Η επιμέλεια από πλευρά των επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό στην αλυσίδα αυτή εφοδιασμού. Το ΕΛΚ και το ΙΣΕΡ θέλουν να αποκλειστεί υποχρέωση από αυτήν τη ρύθμιση. Ευχαριστούμε. Begin τώρα, κύριε Βεγγίνη, για ένα λεπτό δεν είναι εδώ όμω. οπότε περνάμε τώρα στην κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Η Ευρώπη έχει τη μοναδική ευκαιρία και την ηθική ευθύνη να θέσει τέλος στο εμπόριο μεταλλευμάτων από τέτοιου είδους ε, περιοχές. Οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνε ε, θέλουν ε, οι ίδιες από μόνες τους να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα και θα πρέπει να τις καταστήσουμε υπεύθυνε να συμμετάσχουν από μόνες τους έτσι ώστε να συνεισφέρουν με διαφάνεια και προσήλωση στους στόχους μας. Είναι υποχρέωσή μας να δράσουμε ε, με τρόπο απόλυτο για όλη την αλυσίδα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς. Ε, ε, ο κ. Μουκβέμπε το ζήτησε και του το χρωστάμε. Γιατί αν δεν δράσουμε με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε συνένοχοι μιας βαρβαρότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ροδρίγκες Πινιέρο Φερνάντες τώρα. Δεν τη βλέπω όμως στην αίθουσα. Οπότε το λόγο έχει τώρα η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Παρακαλώ. Πέρσι χειροκροτήσαμε τον κύριο Μακβέμπε όρθιοι εδώ πέρα πολλές φορές για την ακούραστη προσπάθειά του να φροντίζει τα παιδιά και τις γυναίκες που είναι τα πραγματικά θύματα αυτού του εμπορίου. Ε, ζητήσαμε ε, ζήτησε ε, τη δράση ε, υποχρεωτικής εφαρμογής, δεσμευτική δράση και αυτό κάναμε και αυτή τη φορά. Ήταν ανεπαρκής μέχρι τώρα νομοθεσία περί της επαρκούς επιμέλειας του due diligence και χρειάζεται πιο ισχυρή δράση. Ψηφίσαμε δεσμευτικές, δεσμευτικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνηση τέτοιων μεταλλευμάτων. Ε, ψήφισα υπέρ προκειμένου να δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα περσινά χειροκροτήματα ε, με ανθρωπιστική δράση σε αυτή την περιοχή εξόρισης μεταλλευμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Στάλτον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εμείς ε, ε, δεν θέλουμε να υπάρχει ένοπλη σύραξη ανάμεσα σε συγκρόμους πλευρές, αλλά εγώ δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την έκθεση, διότι θέλησα να επιβάλλουν κάποιο σύστημα. Εγώ ε, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να υπάρχει ένα εθελοντικό σύστημα, γιατί ένα υποχρεωτικό ε, θα ζημιώσει την οικονομία χάρη, υπάρχουν περιοχές ε, όπου η εξόριξη είναι η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να υπάρξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι αποφεύγουν κάποιες περιοχές. Έχουμε φτωχές περιοχές, ε, όπου δεν μπορούν να υπάρχουν υπεύθυνα προγράμματα και αυτό υποσκάπτει όλη αυτή την ιδέα της νομοθεσίας. Είναι κακή νομοθεσία, δεν θα αντιμετωπίσει τα καυτά θέματα, απλά θα τιμωρήσει τους πιο φτωχούς λαούς στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης ε, αυτής γιατί ε, και ιδιαίτερα μέσα τροπολογίες όπως η 154, 155, ε, δεδομένου ότι αυτές ε, προβλέπουν ένα σύστημα υποχρεωτικής εφαρμογής. Η, η υπεύθυνη προμήθεια μεταλλευμάτων από περιοχές συγκρούσεων είναι πάρα πολύ σημαντική δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές τέτοιων μεταλλευμάτων οι εξαγωγέ αυτών των μεταλλευμάτων από ένοπλες ομάδες ε, που ε, χρηματοδοτούν πολύ συχνά ένοπλες συγκρούσεις με τεράστιες τρα, τραγικές συνέπειες στον ε, πληθυσμό είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν. η Κομισιόν, οι προτάσεις της Κομισιόν δεν ήταν αρκετές. Ε, συγγνώμη, της Επιτροπής δεν ήταν αρκετές. Γι' αυτό το λόγο ε, προτείναμε πιο ε, αυστηρές τροπολογίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα κομμάτια της αλυσίδας και συμπεριλαμβανομένων όνων των μεταλλευμάτων που προέρχονται από ζώνες σύγκρουσης. Πολύ ωραία και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για την άδεια μητρότητα πρώτη παρέμβαση. Κυρία Σόιντροβα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εξηγήσω γιατί κράτησα θέση αποχής στην τελική ψηφοφορία και δεν στήριξα το τελικό κείμενο. Νομίζω ότι για να στηρίξουμε τις γυναίκες στην άδεια μητρότητας και να έχουμε καλύτερες συνθήκες προκειμένου να είναι συμβατός ο ρόλος τους ως ε, γυναίκες στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή είναι κάτι πολύ βασικό και είναι προς το συμφέρον των χωρών μελών. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν με το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο για την υποχρεωτική άδεια πατρότητας. Νομίζω ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συμφωνήσουν. Το σχέδιο ψηφίσματος ζητάει επίσης να επανέλθουμε στο παλιό σχέδιο οδηγία που 7 χρόνια διαπραγματευόμαστε. Πρόκειται για ένα διέξοδο στο οποίο έχουμε φτάσει. Γι' αυτό και προτιμάω να στηρίξω τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποσχέθηκε η Επίτροπος Βερέιβα. Ευχαριστούμε ο κύριος Πετήρα, ένα λεπτό. Ή κυρία Πετήρ, συγγνώμη. Ο, ο κύριος Πετήρ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την πρόταση για την άδεια μητρότητας. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως και επιθυμώ οι γυναίκες να εξασφαλίζονται στον κόσμο της εργασίας και υπάρχουν από αυτού πάρα πολλοί κανόνες. Το θέμα της ε, προστασίας μητρότητας στην Πολωνία μου ρυθμίζεται διαφορετικά από ότι στην Μάλτα, στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει δηλαδή σχέση με κοινωνικούς πολιτισμούς και κοινωνική ευθύνη των ε, κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν πρέπει να υπάρχει διαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτών. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και γι' αυτό εγώ καταψήφισα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κλούν, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Η κυρία Κλούν. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο θέμα της πατρικής άδειας και οι πατεράδε θα πρέπει να μπορούν να μείνουν στο σπίτι και εμεί θα πρέπει να του βοηθήσουμε για να μοιράζονται τι ευθύνε για τα καινούργια παιδιά. Δεν πρέπει οι ευθύνε να βαρύνουν μόνο τι γυναίκε. Θα πρέπει να εισαχθούν και καλύτερα κανόνε για την πατρική άδεια. Ιδιαίτερα όταν θέλουν να αφήσουν για λίγο την καριέρα του. Η, η πατρική άδεια θα εξασφαλίσει καλύτερη ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, φοβούνται μήπως χάνουν και τους άνδρες εκτός από τις γυναίκες. Θα πρέπει να αλλάξουν αυτή την άποψη και το κράτος θα πρέπει να τους βοηθήσει. Ασφαλώ και αποτελεί κόστο για τι επιχειρήσει η απουσία ενό εργαζομένου, αλλά θα πρέπει και οι επιχειρήσει να το δεχτούν ότι, ως ένα ακόμα από τα πάγια κόστη των επιχειρήσεών τους υπάρχουν οικογένειες που ε, δεν μπορούν με άλλο τρόπο να αποκτήσουν παιδιά και δεν είναι δυνατόν να μην αποκτούν παιδιά επειδή θα κοστίσει κάτι λίγο στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται οι γονείς. Ο πρόεδρος διακόπτη. Δεν βλέπω την κυρία Μλίναρ. Περνάμε στην επόμενη μιλήτρια που είναι η κυρία Γκίλ για ένα λεπτό. Ψήφισα υπέρ γιατί είναι απαράδεκτο να μπλοκάρετε ακόμα ε, το θέμα της άδειας μητρότητας στο Συμβούλιο και μάλιστα ακούγονται οι φήμες ότι μπορεί να ε, αποσυρθεί και η πρόταση ως κομμάτι της, του, ε, του προγράμματος REFIT. Ασφαλώς και χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική νομοθεσία στην Ευρώπη, ε, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θέματα όπως η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας που επίσης συνδέεται, δεν ε, θεωρούνται ως ε, θέματα κλειδιά ε, για τα οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει προσπάθεια. Το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και τέτοιου είδου θέματα που επηρεάζουν όλη την κοινωνία δεν είναι δυνατόν να η δράση μας να στηρίζεται σε οδηγίες του 1992 που δεν ε, είναι προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα. Πάνω το 50% ε, των ημερών των γυναικών ε, στη χώρα μου εξαρτάται από τέτοιου αντισμητρότητας. Θα πρέπει η Κομισιόν να βρει μια λύση και όχι να διαλέξει την εύκολη λύση του να πετάξει στο κάτω των απορριμμάτων αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φλάνναγκαν. Κοιτάξτε, εγώ υπερψήφισα διότι πιστεύω ότι αυτό είναι και το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς ε, από την Ολλανδία προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπου μπορέσαμε να αποκτήσουμε περισσότερα δικαιώματα παλαιότερα. Τώρα μας φαίνεται ότι υπαναχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως όσον αφορά την άδεια, ε, τη γονική άδεια, αποφασίσαμε γυναίκα μου και εγώ να αποκτήσουμε μωράκι και αποφασίσαμε να μείνω εγώ στο σπίτι να το προσέχω. Και έπρεπε να αντιμετωπίσω τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πρώτο που μπορεί να κάνει αυτός ο θεσμός, αν κάτι λείπει για την άδεια μητρότητας ή πατρότητα να μην λέτε ότι δεν μας ενδιαφέρει ε, και ότι όσοι ε, κάνουν χρήση αυτού είναι απλά τεμπέλιδες. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποιος ενδιαφέρεται για το μωράκι και θέλει να μείνει σπίτι να το προσέχει. Δεν πρέπει λοιπόν να αποδίδετε τέτοιους χαρακτηρισμούς για κάποιους που προσπαθούν να κάνουν το σωστό πράγμα. Και αυτό ισχύει κυρίως ε, ε, για τις ε, γυναίκες δημοσιογράφους, κάτι που είναι και πολύ παράδοξο. Τώρα κυρία Πετήρ, ευχαριστώ. Λυπάμαι πολύ γιατί η οδηγία για την άδεια μητρότητος προτίθηκε από τα 90 και βρέθηκε σαν διέξοδο στο Συμβούλιο και λυπούμε που δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία. Στις περισσότερες χώρες μέλη ήδη υπάρχουν διάφορες διατάξεις και μερικές φορές καλύτερες από αυτές που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Κράτησα θέση αποχής κατά την ψηφοφορία γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται νέες προτάσεις. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες που πρέπει να διασφαλίσουν ότι και οι μητέρες και οι πατεράδες μπορούν να κάθονται με τα παιδιά τους τους πρώτους μήνες ή τα πρώτα χρόνια ζωής τους. Χρειάζεται λοιπόν νομοθεσία που θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν στους εργαζόμενους τους τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά και να μένουν με τα παιδιά τους στον πρώτο καιρό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Σίλβια Κώστα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το ψήφισμα αφορά σε κάτι στο οποίο έχουμε ήδη, ε, για το οποίο έχουμε ήδη αποφασίσει από το 1992, να έχουμε δηλαδή άδεια μικρότητας. Δεν έχει νόημα για την απόφαση αυτή να την παίρνουν τα κράτη-μέλη προσπάθεια είναι να μεριμνήσουμε για την ευημερία ε, της μητέρας, του πατέρα και του παιδιού. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στις 14 εβδομάδες στην οδηγία του 92. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα για να λάβουμε υπόψη την υγεία των μητέρων και των παιδιών. Και σε περίπτωση οικονομικής κρίσης ή κρίσης απασχόλησης, σε περίπτωση φτώχειας, να επιτρέψουμε στις γυναίκες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει σήμερα λοιπόν να τους προσφέρουμε και άλλες ευκαιρίες και να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις. Επομένως, ε, πρέπει να είναι πιο εύκολη η δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλο και περισσότερες γυναίκες. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και η επόμενη ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου θα πρέπει να επανεξετάσει τις νομοθετικές διατάξεις. Μετά από δύο θητείες δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να υπάρχει μια οδηγία που δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Κώστα. Τώρα θα ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για ε, τα ε, δικαιώματα των αναπήρων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Κώσα από πλευράς ΕΛΚ είναι ο πρώτος ομιλητής. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Η κυρία Κώσα μάλλον. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δούμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση για όλα όσα προτάθηκαν στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τις εξή ε, παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Καταρχάς, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να συμμετάσχουν. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες ε, που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την συμφωνία αυτή. Μία δεύτερη παρατήρηση τώρα. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κληθεί. Άλλωστε αυτό το απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπάρξει διάλογος με τον ΟΗΑ για το θέμα αυτό. Κατά τρίτον, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει πραγματικά το πακέτο αυτό να δημιουργήσει μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια για όλο τον κόσμο το συντομότερο δυνατόν. Και χρειαζόμαστε λοιπόν τις ε, σχετικές, ε, το συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά και τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αυτού του πακέτου. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι εδώ λαμβάνει η χώρα μια παρακολούθηση και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι επιτροπές ε, ΕΜΠΛΕ, ΛΥΜΠΕ και άλλες επιτροπές πάντα το υποδεικνύουν αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει και μια συμβολική σημασία για όλους μας. Χαίρομαι που συνεργαστήκαμε επικοδομητικά στην ομάδα και θέλω να συνεργαστούμε και στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος Πόσπης έχει το λόγο. Δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Ως εκ τούτου θα περάσουμε στην κυρία Σόιντροβα.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 στην πρωτοκαθεδρία και να δίνει το καλό παράδειγμα. Και γι' αυτό λοιπόν το υπερψήφισα και σέβομαι ιδιαίτερα τον, την εμπλοκή, τη δέσμευση των συναδέλφων. Ο προκάτοχος μου, ο κύριος ε, Κόσα είναι ένας από τους ενεργούς φορεί τον τομέα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δραστηριοποιείται όσο θα έπρεπε. Ακόμα και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απασχολούν επαρκή αριθμό ατόμων με αναπηρία. Η κριτική δε που ακούμε ξέρω ότι δεν ε, μας ικανοποιεί. Αλλά δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρόεδρο Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκίλ. Για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στήριξα αυτή την πρόταση ψηφίσματο γιατί περισσότερα, πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίε και όσοι του φροντίζουν έχουν τι ίδιε ευκαιρίε με όλου του υπόλοιπου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίε ε, ζουν και θέλουν να δουλέψουν. Το μισό του 1,3 εκατομμυρίων έχει δουλειά. Λιγότερο από ένα τέταρτο εξ αυτών έχουν προσόντα και όσοι του φροντίζουν είναι σε εξίσου κακή κατάσταση κατάσταση γιατί το 85% δείχνει και λέει ότι το να βρει κανεί σωστή φροντίδα για τα παιδιά που έχει τα οποία είναι ανάπηρα είναι τεράστιο εμπόδιο στην καριέρα του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 700.000 παιδιά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν αναπηρίες και οι οικογένειε τους δεν έχουν επιλογές, δεν έχουν αρκετές επιλογές γιατί δεν έχουν ε, ε, κρατική φροντίδα μέρημνα για τα παιδιά που να ταιριάζει στι ανάγκε του. και γι' αυτό θα πρέπει να επιταχύνουμε για να εφαρμόσουμε σωστά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών με Αναπηρίες. Και αυτό είναι καθοριστικό. Ε, το δικό μας κοινοβούλιο πρέπει αυτό να το πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Σενάλοβα παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. 80 εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως και άλλοι πολίτες θα έπρεπε να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Κάτι όμως που δεν ισχύει στην πράξη και τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε όπως είναι η πρόσβαση στην περίθαλψη υγείας, στην αγορά εργασίας, στη στέγαση, στην παιδεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα έπρεπε να προσπαθήσει να εξαλείψει όλα αυτά τα εμπόδια και του φραγμού και να εφαρμόσουμε τι αρχέ του ΟΗΕ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την πράξη της προσβασιμότητας η οποία θα τονίζει και τις συστάσεις του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η σύμβαση τονίζει μόνο τα ελάχιστα, τις ελάχιστες προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να ανυψώσει τις προδιαγραφές και γι' αυτό υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και τώρα έχετε εσείς το λόγο. Είμαι υπέρ αυτού διότι πιστεύω ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι επωφελές μόνο για αυτούς που έχουν την αναπηρία, αλλά για όλους μας. Διότι όλα αυτά που μπορούν να προσφερθούν είναι πολλά. Αν δείτε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια μορφή προβλήματος αναπηρίας. Ίσως να, μην να έχουν αχρωματοψία, αν μην χρησιμοποιήσουν τον υπόλοιπο στο Λονδίνο, το ένα πόδι να είναι κοντύτερο από το άλλο, όλοι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα έπρεπε να αφορά. Προέρχομαι από μια χώρα όπου εδώ και 50 χρόνια οι άνθρωποι έμπαιναν σε ιδρύματα για να κρυφτούν από τις οικογένειες σε περίπτωση που κάποιος θεωρούσε ότι ήσουν η πηγή του κακού και το κακό οδήγησε σε αυτήν την αναπηρία. Είναι υπέροχο σε πολύ κακό κόσμο ότι αυτό είναι κάτι που συνεχώς βελτιώνεται. Και αυτό δίνει ελπίδα. Είμαι 100% υπέρ αυτού, όχι μόνο για τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά διότι πιστεύω ότι είναι εποφελές ε, για όλους. Ευχαριστώ. Κύριε Φλάναγκαλ, συνάδελφε Κλούνε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τα χαράς ε, υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρη συμμετοχή και ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτό πρέπει να προωθείται σύμφωνα με την προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση τα προβλήματα και έχουμε και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα Ανθρώπων αναπηρία και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στατηγική για την Αναπηρία που βασίζεται στη Σύμβαση αυτή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες. Θα πρέπει να τονίσουμε την προσβασιμότητα, έχει προτεραιότητα ε, πρόσβαση σε υπηρεσίες, να υπάρχει πρόσβαση για ανθρώπους με αναπηρία και να προωθηθεί ε, η πώληση μηχανημάτων υποβοήθησης ε, θα είναι πολύ υποφελές για ανθρώπους με αναπηρία αυτό. Στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με αναπηρία που εργάζονται στην ελεύθερη αγορά εργασίας και θα πρέπει να προωθήσουμε και μια, ε, και μια παιδεία που εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους με την αναπηρία και στη διαβίωση εκμάθηση το ίδιο. Ε, έχουμε, έχει ξεκινήσει πρωτοβουλίες για άτομα με αναπηρία, για εκπαίδευση ε, παιδεία, μελέτη για θέματα αναπηρία και διαβίου εκμάθηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά θα πρέπει και εμεί να τα προωθούμε και να τα υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μαριάννα Πέττη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπορεί να εξασκεί τα βασικά ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτικά του δικαιώματα και η αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου θα πρέπει να διαφυλάσσεται. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακριτικές μεταχειρήσεις και δεν θα πρέπει οι αναπηρίες να εμποδίζουν το άτομο να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν υποστήριξα πλήρως και απόλυτα το ψήφισμα αυτό. 80... 18 εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν με αναπηρία στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν την καθημερινή του ζωή ακόμη και σήμερα εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να καταργήσουμε τα προσκόμματα αυτά. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόσουν ε, την ε, Σύμφωνια για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία. Και αυτή η στρατηγική θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες ε, τις χώρες, σε όλα τα προγράμματα. Θα πρέπει τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες σε ό,τι αφορά την οικονομική, πολιτική, κοινωνική του ζωή. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβια Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζουν σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι με κάποιο μορφή αναπηρία, σοβαρή μορφή, ήπια μορφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΙΕ, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία, έχουν επικυρώσει τη σύμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι από όλα τα κράτη-μέλη. Λείπουν ακόμα τα κράτη-μέλη όσον αφορά την επικύρωση συμβάσεω. Όμω είναι σημείο αναφορά απόλυτο, διότι εγγυάται την αναγνώριση τη καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να εντάσσονται πλήρω τα άτομα με αναπηρία ανευθιακρίσεω. Όμως υπάρχουν λήψεις στοιχείων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση στην απασχόληση και όσον αφορά τα δικαιώματα ε, επικότητας. Υπερψήφισα διότι πιστεύω ότι το ψήφισμα κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδου. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει ένα πακέτο για τα άτομα με αναπηρία με στοχευμένε πολιτικέ, ούτω ώστε να υπάρχει μια γραμμή του προπολογισμού συγκεκριμένη για αυτό το σκοπό, αλλά δίνει τη διαθεσιμότητα όπω σαν πρόεδρο Επιτροπή Πολιτισμού να συνεργάζομαι με άλλε επιτροπέ για το θέμα τη ε, της ένταξης των ανθρώπων απειρία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και ζητάμε μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων ενώσεων των εποπτικών της συμβάσεως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Κυρία Ιβάνα Μάλετιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να έχουν ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. Θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για να εργάζονται και να εκπαιδεύονται και για να έχουν ποιοτική ζωή. Όμως στις καθημερινές ζωές αυτών των ανθρώπων αντιμετωπίζουν ε, πάρα πολλά προβλήματα και φραγμούς. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ολιστική επισκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινώντας από την περίθαλψη υγείας, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την συμμετοχή τους στην πλήρη στην κοινωνία και τις καθημερινές δραστηριότητες εντός των οικογενειών τους. Για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε την πρόοδο. Η κοινωνική ένταξη είναι ένας από τους στόχους της ε, Στατηγικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν μπορεί να επιτευχθεί από μόνη της χωρίς προσπάθειες που θα καταβληθούν από όλους τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη. Στην Κροατία 520.000 άτομα υπάρχουν με αναπηρία ε, ε, που έχουν πληγεί σκληρά από την κρίση και από τα μέτρα λιτότητας. Κάποια μικρή πρόοδο έχει επιτεθεί πρόσφατα με την εισαγωγή ποσοστώσεων όσον αφορά την απασχόληση, όμω υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η ζωή του. Το ψήφισμα είναι ελκυστικό, μάλιστα καλεί όλου να εργαστούν ε, για την ευαισθητοποίηση των προβλημάτων των ανθρώπων αυτών και γι' αυτό υποστήριξα αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Πάμε στι επεξηγήσει ψήφου όσον αφορά το ψήφισμα που αφορά την ξυλέλα Φαστιζιόζα. Αυτό... Η κυρία Ρόζα Νταμάτο έχει πρώτη το λόγο εκ μέρους του EFTD για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να συγχαρώ τους συναδέλφους, διότι ψηφίστε και μια πρόταση ψηφίσματος η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με την εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και διερωτώ με ποιο είναι το, ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Εργαστήκαμε ψηρά ημερών για να επιβεβαιώσουμε τις ίδιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώ ε, συμφωνούμε όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου για τι αγωγέ. συμφωνούμε απόλυτα για τη βοήθεια που θα δοθεί στου ε, αγρότε και στην έρευνα, αλλά στο ψήφισμα δεν αναφέρεται καθόλου ανάγκη αναλύσεω κόστου ωφέλου, που μακροπρόθεσμα θα αφορά την στρατηγική ε, κρίση του προβλήματο. Καμία βούληση να επανεξεταστούν τα μέτρα που προτείνονται υπό το φω των επιστημονικών στοιχείων ε, που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα από πολλά μέρη. Αναφέρομαι στην εξαίρεση των φυτών που θα μπορούν να φιλοξενούν την ξυλέλα και των αμπελιών ε, και τις ζημιές ε, που προχαλούνται από τη μεγάλη κλίμακος χρήση φυτοφαρμάκων. Θα μπορούσαμε να εξοδοθεύσουμε έτσι και η γη ε, δέντρα σε μια ακτίνα 100 μέτρων από τα στενές δέντρο. Και επηρεάζονται όλα τα είδη μόνο γιατί ίσως ενδεχομένως να έχουν αυτό το το πρόβλημα. Είναι μειοπικά τα μέτρα και σίγουρα θα έχουν συνέπειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουν κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ και οικονομικέ συνέπειε. Η δική μου η πρόβλεψη δυστυχώς μέχρι τώρα ήταν εύκολη. Ε, όπως μου προτάθηκε από τον κεφαλής του γραφείου σε πρόσφατη συνάντηση που είχα μαζί του, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις προσπάθειες και τις φωνές μας με τις βασικές οργανώσεις των γεωργών και των προσφυστών του περιβάλλοντος και των Ιταλών και Ευρωπαίων, την Φέντερ Bio, την Copagni, την CIA, την Pan Europe αναφέρω και θα θέλουμε να έχουμε ένα έγγραφο τοποθέτησης κοινού θα το παρουσιάσουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναλλακτικέ λύσει που υποστηρίζουμε, που στηρίζονται και από τι ευρωπαϊκέ οδηγίε και που έχουν εγκριθεί από διάφορε φορεί των πανεπιστημίων και των επιστημόνων. Λοιπόν, αμφιβάλλω ότι οι αρμόδιε αρχέ μπορούν ε, να εθελοτυφλούν και να μην επομιστούν τι ευθύνε του μετά από όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταμάτο. Κύριος Μάσιμο Παολούτσι, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι γεές μας στο, και στο Σαλέτο έχουν πληγεί οι γεωργοί μας από την επιδημία που οι κανόνες ευρωπαϊκοί και τα μέτρα τα ευρωπαϊκά δεν μπόρεσαν να ελέγξουν την επιδημία αυτή. Οι γεωργοί μας είναι θύματα και δεν είναι ένοχοι. Οι, ε, οι δεν είναι μόνο βασική πηγή πώληση, αλλά ε, δίνουν και μια ταυτότητα στο τοπίο. Η Πούλια, το Σαλέντο ε, χωρίς τα μεγάλα ελαιόδεντρα που έχουν ηλικία αιώνων θα είναι το Παρίσι σαν να μην έχει τον πύργο του Άιφελ. Είναι καλή η απόφαση που πήρε η Επιτροπή για, για τα φυτογενομικά να μην συνεχιστεί η τρελή ιδέα να εκριζωθούν ε, χιλιάδε δέντρα από τις πληγήσει περιοχές. Αυτό δεν αρκεί, χρειάζονται παρεμβάσεις τουλάχιστον τρει, Πρώτα απ' όλα με τον ορίζοντα 2020 θα πρέπει να τεθούν πόροι για τι επιστημονικέ γνώσει και την έρευνα θα επιτρέψει να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια που είναι ελάχιστα γνωστή. Δεύτερον, χρειάζονται κατεπίγοντα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποζημιωθούν οι ζημιέ που έχουν υποστεί οι διάφοροι γεωργοί και οι σχετικοί φορεί. Και τρίτον, χρειάζεται λογική διαχείριση τη ελεγχόμενη περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Παλούτσι. Ο κύριο Γιάρ δεν είναι εδώ στην αίθουσα. Το λόγο Έχετε κύριε Νότι Μαριά. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα που κατέθεσα από κοινού με άλλους συναδέλφους για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστροφικών αποτελεσμάτων του βακτηρίου της ξυλέλια Φαστιντιώσα. Το ψήφισμα εγκρίνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και ζητά πρώτον να υπάρξει οικονομική στήριξη των έλαιοπαραγωγών που πλήττονται από την ξυλέλα δεύτερον να αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης των ελαιοπαραγωγών τρίτον να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης εισαγωγής φυτών από τρίτες χώρες που ευθύνονται για την εξάπλωση της ξυλέλιας στην ευρώπη. η ξυλέλια είναι ένα επικίνδυνο βακτήριο που εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα οι ελαιοπαραγωγοί στην ελλάδα και στη μεσόγειο θα υποστούν τεράστια οικονομική καταστροφή. χαιρετίζουμε λοιπόν την υιοθέτηση του ψηφίσματός μας για την ξυλέλια και καλούμε την ευρωπαϊκή επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίησή του. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Μαριάννα Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ιταλικοί, οι Ιταλοί γεωργοί ε, φοβίζουν και τους ε, γείτονές τους και τους ε, αγρότες της Κροατίας. Φοβούνται περισσότερο την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών. Στηρίζω αυτό το ψήφισμα γιατί μας προειδοποιεί για τις τρομακτικές συνέπειες τις οποίες ε, αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί, αγρότες γενικότερα. Και χαίρομαι διότι οθετήθηκαν οι προτάσεις μου ως προς την διάδοση της πληροφόρησης ε, που θα πρέπει να γίνεται και τη λήψη προληπτικών μέτρων, μέτρων παρακολούθησης μεταξύ άλλων. Τα μέτρα αντιστάθμισης, αποζημίωσης δεν θα πρέπει να ξεχαστούν γιατί μια ανεπαρκής αποζημίωση θα οδηγήσει σε αντίσταση στην εφαρμογή των μέτρων και αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα τότε ε, θα ε, ε, διαδοθεί ακόμα περισσότερο αυτή η πληγή της ξυλέλαφας στην Διώσα. Οι αγρότες μας θέλουν γρήγορες και σαφείς απαντήσεις. Θα πρέπει να είναι σωστή και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των αγροτών και των ε, ε, ε, επισήμων αρχών. Ευχαριστώ. Ελοκληρώθηκε η για αυτό το θέμα.